Bueno, a ver, tomen asiento todos. Καθίστε παρακαλώ γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. A ver, un poquito de calma. Bueno, a ver, buenos días, buenas tardes. Καλό απόγευμα για όλους. Παρακαλώ λίγη γαλήνη στην αίθουσα. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και δεν έχω και φωνή σήμερα. Δεν θα αρχίσω να σφυροκοπώ τώρα. Σημείο 1 της ημέρησης διάταξης που είναι η έγκριση της ίδιας αυτής της ημέρησης διάταξης. Μικρόφωνο. Ετήσι του κυρίου Ριβελίνη η ψηφοφορία που είναι πολύ σύντομη, δύο τροπολογίες μονάχα. Και η συζήτηση αυτή για το πέμπτο σημείο θα γίνει πριν από την έκθεση της κυρίας Πατράης. Δέχεστε την ημερήσια διάταξη όπως έχει τροποποιηθεί. Ναι. Εάν έχει έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίασή μας θα διαδικτυωθεί, θα μεταδίδεται δηλαδή από τα ρεύματα του διαδικτύου. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι τα πρακτικά της 3 <clears throat> και 4, 3 και 4 και 23 Νοεμβρίου του 2009. Στην περίπτωση που, θα που δεν θα παρουσιαστεί καμία απολύτως ένσταση θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Σημείο 3 της ημέρης διάταξης και εδώ Να σας υπογραμμίσω εδώ ότι έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο η Πιλάρ Χουάρες, μια ε, υπάλληλος Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεισμό της ΑΙΤΙΣ και θα ήθελα να κρατήσουμε ένα λεπτό συγγύης γιατί η Πιλάρ Χουάρες, όχι, όχι μια στιγμή, ξεκίνησε σαν βουλευτής στην Επιτροπή Γεωργίας και Αλληλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαν, βουλευτή, σαν βοηθός του Κολίνο Σαλαμάνκα, ενός ε, γνωστού Ισπανού βουλευτή. Ασχολήθηκε πολύ και με την ε, Γεωργία και με την Αλία, ιδίως η Γεωργία. Πολλοί από εσά ίσως τη γνώρισαν και στη συνέχεια πέρασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ανάπτυξη και Συνεργασία, Νικαράγουα και μετά ΑΕΤ. Ήταν ένα ιδιαίτερα φιλές άτομο και γι' αυτό σας ζητώ να κρατήσετε ενός λεπτού Bueno, a continuación pasamos al Σημείο 5 της ημερησίας διάταξης, έκθεση Ριβελίνη για την ε, συμφωνία της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια περιφερειακή οργάνωση Αλίας και αυτό το θέμα το έχουμε ήδη συζητήσει στο παρελθόν σε διάφορες συνεδριάσεις. Ο κύριος Ριβελίνη έχει συντάξει μια έκθεση με κάποιες τροπολογίες και νομίζω μπορεί να σας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Λοιπόν, δίνω κατευθείαν τον λόγο στον κύριο Ριβελίνη. Και θα ψηφίσουμε αμέσως μετά. Ελπίζω ότι έχετε όλη την ε, κάρτα ψηφοφορίας. Κύριε Ριβελίνη, έχετε το λόγο. Grazie, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και εσάς ε, επειδή δεχτήκατε να συζητήσουμε το θέμα και την να ψηφίσουμε την έκθεσή μου λίγο νωρίτερα. Θα ήθελα να σας δώσω για κάποιες εξηγήσει για μια προφορική τροπολογία η οποία προτάθηκε μετά από τη λήξη τη προθεσμία για την παρουσίαση των τροπολογιών για το άρθρο 15 παράγραφος 1 και λέει ότι τα σειρώμενα δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται στη Μεσόγειο θάλασσα βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 σημείο 2 του κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 1967 κάθετος 2006 για τις αλλιευτικές δραστηριότητες παρασυρώμενων δικτύων στα αποθέματα της Μεσογείου θα πρέπει να έχουν μια αναγνωρισμένη δραστηριότητα ε, ανοίγματος ματιού δικτύου από, 400, από 40 συγγνώμη, χιλιοστά και μετά. Ο υπεύθυνο ε, αλίας στη Γαλλία ζήτησε να ε, προστεθεί στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ε, να υπάρχει αναφορά άνοιγμα ματιού τουλάχιστον 50 χιλιοστών ώστε να συμπεριληφθεί και μία από τις συστάσεις του ε, GCPM που υιοθετήθηκε το 2009. Έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες όσον αφορά στην αξιολόγηση της επιλεκτικότητας ε, του, των διαστάσεων των ματιών των παρασυρώμενων δικτυών και ο κανονισμός 1967 κάθετος 2007 στο άρθρο 9 παράγραφος 3 ε, δίνει έγκριση για δύο είδη δικτυών, 40 χιλιοστών ή 50 χιλιοστών, κατόπιν του εύλογου αιτήματο ε, του ε, εφοπλιστή, του πλειοκτήτη. Ε, να διευκρινίσουμε εδώ ότι επιτρέπεται να έχουν επί τους μόνο ένα εκ των δύο ειδών δικτυών. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα λοιπόν στην ψηφοφορία. Εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, θα ήθελα να ψηφίσουμε καταρχάς την προφορική τροπολογία του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ah, <laughs> ah, Πέραση ψηφοφορία. 21 18 eh, ψηφίσαντες, 18 υπέρ, ένας κατά και δύο αποχές, επομένως εγκρίνεται η προφορική τροπολογία. Στη συνέχεια να περάσουμε στην τροπολογία υπαριθμών 1 άρθρο 28, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 eh, ψήφοι υπέρ, δύο αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία 1 του εισηγητού. Και επειδή είναι ψήφος προσανατολισμού, διότι όπως γνωρίζετε Βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο της διαδικασίας συναπόφασης. Πρόκειται για ψήφο προσανατολισμού και επομένως δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ψηφοφορία αυτή και να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης ψηφοφορία για την πράσινη βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής η συγχύτρια η κυρία Πατράου ο κύριος Λεβίν η κυρία Λεβίν, κυρία Λεβίν. Ναι, Προτείνω να κάνουμε δεκάλεπτη διακοπή μετά την ψηφοφορία, πριν την τελική ψηφοφορία δηλαδή, για να αποφασίσουμε αν τελικά θα υπερψηφίσουμε ή θα καταψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης. Bien. Alguna... Εντάξει. Άλλη παρέμβαση. Κύριε Χιούτον, υποστηρίζω την πρόταση Τη ε, κυρίας εξεβονίμων μου, αλλά θέλω να προτείνω επίσης, επειδή είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία για την κοινή αλληλευτική πολιτική, Βλέπω ότι είναι εκπληκτικό και όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικό ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε στην Επιτροπή μας τα θέματα αυτά μετά από την ε, δημοσίευση της έκθεσης της, έκθεσης, της εισηγήτριας και ελάχιστο χρόνο για να συζητήσουμε τις 420 και 3 τροπολογίες ενώπιον μας. Ελπίζω ότι δεν θα δουλέψουμε με τέτοιο χρονοδιάγραμμα όταν φτάσουμε σε νομοθετικό επίπεδο για το ζήτημα αυτό. Εγώ θα χαιρέτησα ιδιαίτερα την ευκαιρία να παρουσιάσω ενώπιον της Επιτροπής μας τους ε, λόγους που με οδήγησαν να καταθέσω ορισμένες τροπολογίες και ίσως δεν είμαι ο μόνος που θα ήθελα να πράξει κάτι τέτοιο. Κυρία Πατράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο, ούτως ώστε μεταξύ των συναδέλφων ακόμη μια φορά να υπογραμμίσω ότι να υπενθυμίσω μόνο τις προθεσμίες που έχουμε και οι οποίες απορρέουν από τις προθεσμίες με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θυμούνται οι συναδέλφοι ότι ήδη δύο φορές εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή μας ε, προέκυψε αυτό το χρονικό ζήτημα και αρκετά νωρί εξάλλου. Διότι δεν γνωρίζαμε εμεί το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο έπρεπε να κινηθούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η πράσινη βίβλος έχει ανοίξει είχε ανοίξει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου για, άλλες, για διαβούλευση και στη συνέχεια έπρεπε να κάνει τη σύνθεση, τη σύνοψη η Επιτροπή που θα παρουσιαστεί στις αρχές Μαρτίου. Οπότε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν αρκετά σοβαρό αν τελικά δεν εκδίδαμε, δεν δημοσιεύαμε την έκθεσή μας πριν αναλάβει αδίποτε πρωτοβουλία στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ούτως ή άλλως θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία θα ήταν ακόμη σοβαρότερο. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι το θέμα του διαθέσιμου χρόνου έχει συζητηθεί δις και είναι επιζήμιο και για μας και για τους ασυγητές και για τους σκιώδεις ασυγητές. Και παρότι δεν έχουμε ε, αρκετό χρόνο για δουλειά τέτοια εμβέλειας, παρόλα αυτά ακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στο πρόγραμμα της Επιτροπής. Εγώ δύο-τρεις φορές έχω συναντηθεί με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Έχω κάνει λοιπόν συσκέψεις μαζί τους και γι' αυτό είστε κι εσείς μάρτυρες ότι παρότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, έχουμε καταβάλει όλη η προσπάθεια για να το καταφέρουμε ε, και να έχουμε ένα ισχυρό έρισμα για τις εργασίες μας. Λοιπόν, ανεξαρτήτως του χρόνου εργαστήκαμε ε, πολύ καλά μέσα σε ανοιχτό και διαφανές ε, πνεύμα ε, και σε στενή συνεργασία και εργαστήκαμε, μοχθήσαμε όλοι πολύ, όχι μόνο οι σκιώδεις εισηγητές, έτσι, γιατί υπέβαλαν πολύ, πάρα πολλές τροπολογίες, όλα τα μέλη της Επιτροπής, ε, στην πρώτη και στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων και στην πρώτη παρουσίαση της ε, έκθεσης, ε, έκαναν κάποιες προκατακτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γκάλαχερ. Κυρία Πρόεδρε, εν συντομία, κανείς δεν διαφυσμητεί το γεγονός ότι οι εισηγήτρια και οι ισχύοδες εισηγητές, γνωρίζω από τη δική μου περίπτωση της δικής μου ομάδας, ότι έχουν εργαστεί πολύ σκληρά σαν άτομα για να προσπαθήσουν να προχωρήσουν με το θέμα της επεξεργασίας της έκθεσης και της τροπολογίας. Και αν δώσουμε περισσότερο χρόνο ίσως δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Σίγουρα μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση προς τα έξω ότι είναι βεβαιασμένη η διαδικασία για την έκθεση αυτή παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες προτάσεις είχαν διατυπωθεί μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου και ενδεχομένω θα πρέπει να επανέλθει η επιστροφή μας. Εμείς δεν μπορούμε εύκολα να το εξηγήσουμε αυτό σε όλους τους αλείς και στις οργανώσεις των παραγωγών ότι όλα έγιναν χωρίς να εμφανιστούν στην πραγματικότητα. Η δουλειά έγινε μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και της εισηγήτριας. Αυτό διαφέρεται όμως και από τον αριθμό των συμβαστικών τροπολογιών που έχουν διατυπωθεί. Πάντως δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση να δαπανίσουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Ίσως αυτή η έκθεση προχώρησε πιο γρήγορα από άλλες εκθέσεις ίσως σημασία γιατί εγώ τολμώ να πω ότι αυτή η έκθεση θα είναι η πιο σημαντική έκθεση που θα αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος, ε, η κυρία Ρόμπουστ. Κυρία Πρόεδρε, θα, θέλω να, θα ήθελα να εκφραστώ εναντίον των δύο αυτών ε, προλαλήσαντων. Νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Πατράου Νέβες για την εργασία της. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά όλοι μέχρι την τελευταία στιγμή με τις ε, συνεργάτησές της και με τους συντονιστές εργαζόταν η συγγήτρια. Όλοι ασχολήθηκαν με αυτή την έκθεση. Εγώ νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι μια καλή έκθεση και φαίνεται αυτό άμα το δούμε. Τελικά είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα πιστεύω και μπορούμε να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι έχουμε εργαστεί πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο δεν, δεν συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσουμε σε κανένα το πόσο γρήγορα καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, επομένω δεν επιδέχεται κριτική η διαδικασία αυτή. Εντάξει, καταγράφω αυτό το οποίο <clears throat> αναφέρατε και τις ε, ενδεγόμενες αυτές επικρίσεις. Πριν φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης θα διακόψουμε για 10 λεπτά. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό το οποίο ζητάτε. Και από τώρα λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεργαστείτε με την Προεδρία γιατί αλλιώς θα περάσουμε όλο το βράδυ να ψηφίσουμε και μάλιστα χωρίς διερμηνία. Λοιπόν, θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 93, άρχεται ψηφοφορία. <coughs> Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της Απορρίπτεται όμως. Ακολουθεί η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ. Ακολουθεί λοιπόν Εφόσον εκπίπτει η τροπολογία 96, περνάμε στην τροπολογία 121, η οποία όμω όχι αποσυρθεί και θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 19 ψήφου κατά. Τροπολογία 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με 19 ψήφους κατά. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ. Η τροπολογία τώρα εκπίπτει το πρώτο τμήμα τη τροπολογία 102 ψηφίζουμε το δεύτερο μόνο τμήμα τη 102. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Και τώρα απορρίπτεται γιατί υπάρχει ισοψηφία 11-11. Δεν γίνεται δεκτό το δεύτερο τμήμα τη 102 κατά συνέπεια. Εκπίπτουν τώρα η τροπολογία 100, η τροπολογία 101 επίσης και θέτω σε ψηφοφορία την 103, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 15 ψήφους θετικές. Τροπολογία 104, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 19 ψήφοι υπέρ. 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 14 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Ψηφίσουμε την τροπολογία 107. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία και απορρίπτεται με 17 ψήφου κατά. Ερχόμαστε στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Εκπίπτει ο εκ τούτου η τροπολογία 108 καθώς και 109. Θέτω σε ψηφοφορία τροπολογία 110. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 15 ψήφους κατά. Στη συνέχεια, η τροπολογία 111 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. ένας σοσιαλιστής παραπάνω, κυρία Ρόμπουστ. Απορρίπτεται ούτως ή άλλως με 18 ψήφους κατά. Δεύτερο... Το δεύτερο τμήμα εκπίπτει, μάλιστα, πολύ σωστά. Μεγάλο το δίκιο σας. Τροπολογία 266, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 19 ψήφους κατά. εκπίπτει η 112 διότι ενεκρίθη η 95 και περνάμε στη συμβαστική υπαριθμών 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 22 ψήφου. επομένως οι τροπολογία 113, 114, 115 και 116 εκπίπτουν. Και περνάμε στην 117 η οποία είναι συμβατή με τη συμβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 117. Πέρας. Εγκρίνεται με 19 ψήφους. 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 10 έναντι 9 και μίσης αποχής. Σε ψηφοφορία η τροπολογία 119 σε δύο τμήματα. Κύριε Χιούτον, κύριε Φερέ, δεν λειτουργεί το μηχάνημά μου, κυρία Πρόεδρε. Κάθεστε κάπου αλλού, δεν πειράζει. Μα τα λέτε λίγο πολύ γρήγορα και δεν προφθαίνω, λέει ο κύριος Φεραίρα. Μα η τροπολογία σας εγκρίθηκε. Κλείνετε την ψηφοφορία πρωτού προλάβουν να ψηφίσουν όλοι. Μα κρίθη η τροπολογία σας. Τι θέλετε τώρα. Ενεκρίθη. 19 ή 118. Ναι. 19. Κερδίσατε κύριε Φερέ, Δεν έχετε πρόβλημα. Αν δεν σας αρέσει το μηχάνημα βρείτε κάποιο άλλο. 119 σε δύο τμήματα. Και άμα πάω πιο γρήγορα πάω πιο αργά αλλά μετά θα μείνουμε εδώ πέρα μέχρι το βράδυ. Δεν έχω πρόβλημα, τα λέω πολύ αργά αν επιμένετε. 119 είναι καλό. Ε, εντάξει. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι και γρήγορη και αργή συγχρόνω. 119. Πρώτο τμήμα. Ψη, ψη, ψήφι υπέρ. Πέρασε ψηφοφορία. Γίνεται δεκτή με 16 ψήφους. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία απορρίπτεται με 9 υπέρ 11 κατά. Η τροπολογία 120, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. 24-0. Ακολουθεί η τροπολογία 120, 122. Συγγνώμη, λέει πρόεδρο, η 122, όχι συμβαστική τροπολογία, 122 πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται 13-11. Συμβιβαστική. Τροπολογία υπαριθμών 5. <clears throat> Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα όλο το κείμενο χωρίς τη λέξη all στα αγγλικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους. Το δεύτερο τμήμα είναι η επίμαχη λέξη all. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 13 ψήφους έναντι 10. Ω εκ τούτου εκπίπτουν οι τροπολογίες 123, 125, 124, 126, 127 όπως και 128. Και μπορούμε να ψηφίσουμε, λέει πρόεδρο, την 128 ως προσθήκη. Όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι δεν είναι συμβατή με την ε, συμβαστική εκπίπτη και 128. Και ψηφίζουμε την 129 αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 16 ψήφους θετικές. Ακολουθούμε την τροπολογία 130 άρχη ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται με 16 ψήφους. 131. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 ψήφους. 132. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 22 ψήφοι θετικές. Εγκρίνεται. Η 133 έχει εκπέσει. Έχει εκπέσει. Περνάμε στην 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Έχει εγκριθεί με 21 ψήφους. Και τώρα υπάρχει μια προφορική τροπολογία για να προσθεθεί κάτι σε αυτήν την τροπολογία. Βλέπετε το κείμενο στους φακέλους σας. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, κύριε Ευελιάν, μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν πρόκειται να τα διαβάσω τώρα όλα αυτά που λέει. Ψηφίζουμε την προσθήκη των πρασίνων. Αν υπάρχει κάποιος όμως ο οποίος αντιτίθεται, πρέπει να το πει τώρα. Εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία. λήξεις. Εγκρίνεται με 20 ψήφους. 135 εκπίπτει, πάμε στην 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται με 17 ψήφους κατά. 137 που είναι τροπολογία διαγραφής Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμό 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους, επομένως εκπίπτουν τροπολογίες 138, 140, 139 αλλά και 141. 141 όχι ψηφίζεται πράγματι. Πέρασε ψηφοφορία. 20 ψήφοι θετικές εγκρίνεται. Ακολουθούμε τις τροπολογίες 142 θέτω σε ψηφοφορία. Πέρας. Ιτάτε και απορρίπτεται με 18 ψήφους κατά. 144. Δεν εκπίπτει, δεν εκπίπτει, όχι. Ψήφισμα είναι 144. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 145. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται. 13-9. 146 με δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία στο πρώτο τμήμα. Πέρας. Δεν γίνεται δεκτό. 14-9. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. ¿Se vota o no se vota? Bueno, se vota. Abro la votación para la segunda parte. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε τι τροπολογίε 146. Άρχεται η ψηφοφορία, είπαμε. Πέρα. Δεκτή με 15 ψήφου. 147 εκπίπτει 148 επίσης εκπίπτει. 149 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 151. Κατά τμήματα και αυτή. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 14-10. Δεύτερο τμήμα. Θέτω η ψηφοφορία. Λήξεις και αυτό απορρίπτεται 19-4. 152. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 19 ψήφους. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 ψήφοι θετικές εγκρίνεται. Εκπίπτει η τροπολογία 153-154. 155 ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία 155. πέρας. Απορρίπτεται με 15 ψήφους αρνητικές. 156 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους. 157 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται με 15 βότους, ψήφου. ψήφους. τροπολογία 8. Θέτω ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με 21 ψήφους υπέρ. Εκπίπτουν 158 καθώς και 159. Τροπολογία 161. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι. Εγκρίνεται με 22 ψήφους, 162 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι. Εγκρίνεται με 23 ψήφους. 163. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται με 21 ψήφους. 164. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι, Εγκρίνεται με 16 ψήφους. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι, Εγκρίνεται με 23 ψήφους. Εκπίπτει 165 καθώς και 166. Η 10 συμβιβαστική έχει αποσυρθεί. Ψηφίσουμε την 167. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι. Απορρίπτεται με 16 ψήφους κατά. 168. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ. 170 έχει εκπέσει. Διότι είναι εκρήτη 168. 170 εκπίπτει 169. Η 167 μόνο ως προσθήκη στην 169. Η 169. Πέρας. Εγκρίνεται με 19 ψήφους. 172 άρχεται η ψηφοφορία λήξη. Δεκτή με 23 ψήφου. Αποσύρθηκε η συμβαστική 11. Ψηφίσουμε την 173. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 12-10. Ψηφίζουμε τώρα την 226. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 15 ψήφους κατά. 227. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική υπαρτιμό 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με 23 ψήφους, εκπίπτουν ως εκ τούτου 150, 174, 175, 177 και ψηφίζουμε τώρα σαν προσθήκη την 176 με το κείμενο το πρόσθετο που αναφέρεται στο κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία στην 176 ως προσθήκη. Πέρας. Απορρίπτεται με 19 ψήφους κατά. 178. άρχιδη ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται με 17 ψήφους. 179. άρχιδη ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. 180. Άρχιε την ψηφοφορία. Λίγη. Δεκτή. 181. Άρχιε την ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη εγκρίνεται. Εκπίπτουν 182, 184, 185, 183, 186 και 187. Περνάμε στη συμβιβαστική 14. Σε τμήματα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της συμβαστική 14, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξει. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτό. Εκπίπτουν 188, 189, 334 ή 191. Ψηφίσουμε την 190. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ένας του ΕΛΚ παραπάνω βουλευτής ψηφίζει. Κύριε Αντινόρη, Αντινόρο, κάποιος από εσά δεν πρέπει να ψηφίζει. Εντάξει. Φεύγει ο κύριος Μεντεσδεβίγο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας παρόλα αυτά. Πού έχουμε μείνει τώρα, τα χάσα. Την 190 την ψηφίσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία στην 190. Εγκρίνεται. 193 και 208 που είναι δίδυμες και ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνονται. 194. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. <clears throat> Δεκτή. 195. Άρχεται. Λήξεις. Δεκτή. 196. Άρχεται. Ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 197. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 198. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. 199. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 200. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται με 15 ψήφους κατά. 201 άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 202 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. 14-9. 203. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται με 13 ψήφους κατά. 204. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 205. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 206. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. 207. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. 209. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται με 18 ψήφους κατά. Συμβιβαστική τροπολογία 15 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται με 24 ψήφους. Εκπίπτουν τροπολογίες 210, 212, 211, 213, 214, 171 και ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 215. Άρχεται η ψηφοφορία. κλείνει. Εγκρίνεται με, 11, με 12-11. Συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι χωριστή ψηφοφορία, συγγνώμη, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμό 16 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Δεκτό, το δεύτερο τμήμα. Εκπίπτουν οι 216 καθώς και οι 220. Ψηφίζουμε 218. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 12-10. Επομένως εκπίπτει 217 Πάμε στην 219. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται 15-9. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται εκπίπτουν οι 2-2-1 και 2-2-2. Περνάμε στις 223 και 224 που ταυτίζονται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 13-9. 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. 228. 2-8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 15 ψήφους. 231. Άρχεται η ψηφοφορία. λήξης απορρίπτεται με 16 ψήφους κατά και 7 υπέρ 2.32 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και αυτή απορρίπτεται με 19 ψήφους κατά. Συμβιβαστική τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε δύο τμήματα, συγγνώμη, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Λήξεις. Και το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα εκπίπτουν οι 230, 229 καθώς και οι 233. Η 230 ψηφίζεται. Άρχεται ψηφοφορία στην 234. Λήξεις. Εγκρίνεται. 2.35. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 2.36 που είναι συμβατή Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. 2.37 σαν προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. 2.38. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι 240, 242, 239, 241. Ψηφίζουμε την 243. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις εγκρίνεται. 2.44 άρχεται. Λήξεις. Απορρίπτεται. κάνει ψήφοι κατά. 2.47 λήξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.48. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται με 14 ψήφους κατά. Δύο Λήξεις. Εγκρίνεται με 19 ψήφους. Εκπίπτει τώρα η 250 όχι, όχι, λέει η γραμματεία. Είναι συμβατές. Συμβατές. 250. Ψηφίζουμε. Άρχεται. Λήξεις. Εγκρίνεται. 251. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 252. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.53. Άρχεται. Λήξεις. Δεκτή. 254. Άρχεται. Λίγεται. Δεκτή. 255. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 ψήφι κατά. 2.56. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 2.57 εξέπεσε. 2.58 ως προσθήκη μόνο. Άρχεται η ψηφοφορία στη 258. Λήξεις. Απορρίπτεται με 14 ψήφους. 2.59. Άρχεται. Λίγοι και λιγότεροι. Εγκρίνεται. 260. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 261 εκπίπτει. 262 εκπίπτει λέει η πρόεδρος όχι, όχι, όχι, όχι δεν έχει εγκριθεί η 259 ναι, εκπίπτει τότε 263 εκπίπτει και 264 είναι συμβατή ψηφίζουμε τη 264 άρχεται η ψηφοφορία λήξεις εγκρίνεται 265. Άρχεται. Λήξεις. Εγκρίνεται. 268. Άρχεται. Λί. Εγκρίνεται. 267 εκπίπτει. 269 είναι συμβατή. Ψηφίζουμε τη 269. Πέρας. Εγκρίνεται. 270. Έχουμε ένα πρόβλημα. 270 άρχεται. Λήξεις. Εγκρίνεται. Η 271 έχει αποσυρθεί. Πάμε στη συμβιβαστική 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εκπίπτουν 272, 276, 273, 275 και 274. Ψηφίζουμε τη 277. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Ε, 278. Άρχεται η ψηφοφορία. λήξης. Απορρίπτεται. 279. αρχεται ληξει Λήξης. Εγκρίνεται 12-11. 280. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξει. Εγκρίνεται με 14 ψήφους. 281. Άρχεται. Λύξεις. απορρίπτεται με 10 κατά. Συμβαστική τροπολογία 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξει. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Λήξει. Εγκρίνεται επίσης εκπίπτουν 282, 283, 285, 284 και 286. Ψηφίζουμε την 287. Άρχεται. Λήξεις. Εγκρίνεται με 14 ψήφους υπέρ. Συμβαστική 22 έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 288. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. 346. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 289. Άρχεται. Λήξεις απορρίπτεται με 15 ψήφους κατά 290 άρχεται λίγη εγκρίνεται με 16 ψήφους 291 σε τμήματα, σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα άρχεται λίγη απορρίπτεται δεύτερο τμήμα άρχεται Λίγη. Απορρίπτεται επίσης. 2.92 και 2.93 που ταυτίζονται. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτονται. 2.95 άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 294. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. 296. Άρχεται. 12.10. 12-10 απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. Αφού εγκρίθηκε. 297. Η 297 καταπίπτει. 299 επίσης. 200... 98, 301, 304, 303, 302, 305 ε, καταπίπτουν. Να περάσουμε λοιπόν στην 300, η οποία είναι συμβατή με το συμβιβασμό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 13 ψήφους. Η 306. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 307. Εγκρίνεται. Άρχεται συγγνώμη ψηφοφορία. Ε, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 308. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 309. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 310. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 14 ψήφους κατά και 9 υπέρ. Η 311 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκαν οι προηγούμενες. 312. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 313. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Γκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ. 314. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 12 ψήφους υπέρ, 10 κατά. 317. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 317. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 318. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Στη συνέχεια. Συμβιβασμός υπαριθμών 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 319, 321, 320, 322. Ψηφίζουμε κατά τμήματα την 323. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται και αυτή. Η 324 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκαν οι 308 και 310. 325, 326 είναι τα φτώσιμες. Ε, τις υποβάλλουμε προς ψήφιση λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 327, οι 328 και η 329. Ο συμβιβασμός 25 αποσύρθηκε. Καταπίπτουν οι 330, 331, 332 και η 333. Και ψηφίζουμε την 335. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η 336, γιατί εγκρίθηκε η 335. 337 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και αυτή εγκρίνεται. Η 338 καταπίπτει. 339. Άρχεται η ψηφοφορία για την 339. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 ψήφοι κατά. 340. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 341 εκπίπτει, 342 επίσης και η 340 είναι συμβατή με την 340. Ψηφίζουμε λοιπόν την 343. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 344. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 345. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 347 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 175. 348 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 349 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 350 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 351. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 352. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 353. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 14 ψήφοι κατά 8 υπέρ μόνο. Ο συμβιβασμός υπαριθμών 26 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 160, 354, 355. Και εκπίπτει επίσης το δεύτερο τμήμα της, της 356. Θα ψηφίσουμε μόνο το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 356. Πέρας ψηφοφορία, Εγκρίνεται. 357. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 358. Τι έπαθε αυτή. Εκπίπτει λοιπόν, περνάμε στον ε, συμβασμό 27, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι 359, 360 και 361. Ψηφίζουμε την 362. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 363 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 364 άρχεται η ψηφοφορία, λήξη, εγκρίνεται. 365 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Η 366 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 367 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 368 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 369 άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ...370. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 371. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 372. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 373. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 375. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 374 ως προσθήκη. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 376 κατά πίπτη και περνάμε σε 377 κατά τμήματα. Uh, Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειαζόμαστε την κατατμήματα ψηφοφορία πλέον, επομένως θα αποσύρουμε το άτομα. Εμείς το είχαμε ζητήσει, δεν μας ε, απαιτείται πλέον. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο της 377. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Αγκρίνεται. 378. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 379. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 380. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 381. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 382 άρχεται. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 420 εκπίπτει. 421 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται καταπίπτει η 2.45 του κ. Φερέιρα και ψηφίζουμε τώρα τον, τη συμβιβαστική τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Καταπίπτει η 246 και η 383. Ψηφίζουμε την 384. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. 422. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 385. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία, Εγκρίνεται. 423. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 386. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 387 αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε την 388. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 389. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 390. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 15 ψήφοι κατά. Ψηφίζουμε τώρα τον συμβιβασμό υπαριθμών 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 391 και 392. Ψηφίζουμε την 393. Άρχεται η ψηφοφορία. Πίπτη. Ε, λήξη. Εγκρίνεται. 11-10 για μία ψήφο. 394. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 395. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 ψήφοι κατά. 396. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 17 ψήφους. 399. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία Απορρίπτεται 15 ψήφοι κατά 6 υπέρ. Ψηφίζουμε τώρα τον συμβασμό 30. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται και αυτό. Εκπίπτουν 397, 398, 400, 401, 402. Και επειδή δεν εγκρίθηκε η 399, ψηφίζουμε την 403. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 404. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 ψήφοι κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν την 405. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 406. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 ψήφοι κατά. 407. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 408. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 409. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 410. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 411. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 412. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 413. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 414. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 415. Άρχεται. Λήξη τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια, συμβιβασμός υπαριθμός 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκπίπτει 416 και ψηφίζουμε την 417. Άρχεται... Α, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Συγγνώμη δεν λειτουργήσε το σύστημα και δεν μπόρεσα να ψηφίσω, αλλά επειδή ούτως ή άλλως την υπερψηφίσαμε, δεν φαίνεται ποιο ψήφισε. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, το λέω γιατί κάποιο πρόβλημα είχε να σημειώσετε την ψήφο μου. 417. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 32 αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν την 418. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 192. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 315 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Η 192 εγκρίθηκε, επομένως το πρώτο τμήμα Καταπίπτει. Και ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 315. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 419. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στα εκτιμώντας. Εκτιμώντας 1. Τροπολογία 1, συγγνώμη. Τροπολογία ε, υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία Εγκρίνεται. 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 15 ψήφους κατά. Η 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 10 ψηφίζεται. Ψηφίζουμε τη 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 12 ψήφου κατά. 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 14 ψήφου κατά. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 16 ψήφου κατά. 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 18. Συμβατή με τη 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Η 19 καταπίπτει. Η 20 είναι συμβατή με τις 17, 18, 19. Άρχεται η ψηφοφορία για την 20. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 15. 21 δεν καταπίπτει. Η 21 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 22 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψήφο. 12-11. Τροπολογία 24 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 10-10 εκπίπτει. Απορρίπτεται εννοεί η πρόεδρος. Και από εκεί και πέρα ε, καταπίπτει το δεύτερο τμήμα γιατί δεν έχει νόημα. Ψηφίζουμε λοιπόν τον 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26 άρχεται ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, εκπίπτει γιατί εγκρίθηκε 25. 27 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 33. Άρχεται η ψηφοφορία για το συμβιβασμό. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 28, 30, 31, 32, 33, 34 και 29. Ψηφίζουμε. Συμβαίνει κάτι, ρωτάει η Πρόεδρος. Όχι. Την 35. Σε φιέρα, perdón, Πέραση ψηφοφορία. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα, λέει η Πρόεδρος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 17 ψήφους κατά. Ψηφίζουμε στη συνέχεια το συμβιβασμό 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 36, 38, 39, 40 και 41. Ψηφίζουμε την τροπολογία 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 19 ψήφους κατά. Στη συνέχεια, συμβιβαστική τροπολογία 35, την οποία ψηφίζουμε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται και αυτό. Εκπίπτουν οι 46, 47, 48, και 50. Εκπίπτει και η 49, η οποία είναι συμβατή. Συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία για τη 49. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 συμβατή ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 58, εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 59 συμβατεί με την 58, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Κατόπιν, περνάμε στην τροπολογία 60, την οποία ψηφίσουμε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της 60, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία 61, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την 66. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και αυτή. Ψηφίζουμε λοιπόν την 67. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 17 ψήφους. 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 14 ψήφους κατά. 71. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 72. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13 ψήφοι υπέρ 10 κατά. 73. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας απορρίπτεται 16 ψήφοι κατά 75 άρχεται η ψηφοφορία λήξη εγκρίνεται 74 κατά τμήματα Συμβατεί με την 75 ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία Πέραση της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται και αυτό με 12 ψήφους υπέρ 9 κατά. Τροπολογία 76. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 77. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 78. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 17 ψήφους κατά. Στην 79 έχουμε και προφορική τροπολογία. Έχετε το κείμενο εδώ. Εάν δεν ε, έχει κάποιο αντίρρηση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται 13 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. 81. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι 84 και οι 85 είναι συμβατοί ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία για την 85. Πέρασε τη ψηφοφορία και εγκρίνεται με 12 ψήφους υπέρ και 9 κατά. Τροπολογία 86. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 87, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 88, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 90, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Τελευταία. Επιτέλους. Άντε. Τα καταφέραμε. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ωραία. Όπως έχουμε συμφωνήσει 10 λεπτά ακριβώς, έτσι στις παρατέταρτο όλοι εδώ να ψηφίσουμε αν έχετε την ευγενή καλοσύνη διότι τα... Ε, πρέπει να βιαστούμε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Καθίστε παρακαλώ. Σοσιαλιστές, μήπως μπορείτε να λύσετε το πηγαδάκι και να καθίσετε. cinco minutos de más sobre los diez que habían sido solicitados. Έχουμε φάει και πέντε λεφτά παραπάνω πέραν των δέκα που είχαμε πει. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Καθίστε όλοι, έχετε την κάρτα σας στη μηχανή ψηφοφορίας. Πάμε λοιπόν, τελική ψηφοφορία. Άρχεται η τελική ψηφοφορία. Σε cierra Λίγη τελική ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Ψήφισαν 24, 15 υπέρ, 9 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Πατράου Νέβες. Bueno, hemos hecho un trabajo, yo creo que bueno. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η εργασία μας και για να συνεχίσουμε είμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. ver, Και συνεχίζουμε στην ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Χάρμ Κώστερ, εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας για τον έλεγχο της σας παρακαλώ, λίγη γαλήνη, λίγη σιωπή, λίγη ησυχία. Μήπως μπορείτε να σιωπήσετε. Αν δεν θέλετε να σιωπήσετε, να βγείτε από την αίθουσα τουλάχιστον. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις υποδομές αυτού του φορέα. Κύριε Αντινόρο, βρε κύριε Αντινόρο, δεν έχω φορεί και να κάνω να φωνάζω για να σας επαναφέρω στην τάξη. Τι είναι αυτό είχαμε προβλέψει να πάει μια αντιπροσωπεία στην εκτελεστική αυτή υπηρεσία στην, στο Βίγο. Ξέρετε ότι υπήρξε πρόβλημα με τις ε, μετακινήσεις αυτής. επειδή είχαμε τις ακροάσεις των επιτρόπων χρειάστηκε να ακυρώσουμε όλα αυτά τα ταξίδια παρά το γεγονός ότι αλλάξανε οι ημερομηνίε για τους επιτρόπους. Στη συνέχεια με τα προβλήματα που είχαμε μπορούμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε μα, λίγο σεβασμό για τον κύριο Κώστερ Έχουμε ζητήσει λοιπόν από τον Διευθυντή του Φορέα για την Αλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει και να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασία που έχουν για το 2010 και τα επιτεύγματά του του 2009 και φυσικά θέματα όπως η παράνομη και ε, μη ρυθμιζόμενη αλία, η άναρχη και παράνομη αλία συγκεκριμένα, όλα αυτά τα οποία κάνει η υπηρεσία ελέγχου για να αντιμετωπίσει διαθέματα, Ξέρετε ποιε είναι οι ευαισθησίε της Επιτροπής μας κύριε Κώστερ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ για το έργο του φορέα σας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός σε ελεκτικό επίπεδο και που έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Σας δίνω το λόγο λοιπόν να εξηγήσετε σε όλους ποιε είναι οι δραστηριότητέ σα και ποιο ήταν ο απολογισμό του 2009. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αλίας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ ε, για την ε, πρόσκληση για να σας παρουσιάσουμε τις ε, δραστηριότητες και το πρόγραμμα εργασιών μας. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τις δραστηριότητες υπηρεσίας. Εδώ και 1,5 χρόνο Έχουμε την έδρα στο Βίγκο, στην Ισπανία. Το 2007 αρχίσαμε πρώτα απ' όλα στις Βρυξέλλες και μετακομίσαμε το 2008 στο Βίγκο. Και τώρα μπορούμε να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας βάσει της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Συντονίζουμε τον έλεγχο και την επιθεώρηση ε, και όλες οι σχετικές δραστηριότητες των κρατών μελών. Έχουμε κοινά προγράμματα ανάπτυξης με συνδυασμό των εθνικών ελεγκτικών πόρων και συντονισμό των επιθεωρήσεων που γίνονται στα κράτη-μέλη. Επίσης, επικουρούμε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Το 2010 ελπίζουμε να επανδρώσουμε με 60 άτομα την υπηρεσία για να επιτελέσουμε αυτά τα καθήκοντα. Θα σας εξηγήσω εν συντομία την αποστολή, τη στρατηγική και τους στόχους της υπηρεσίας, τα προκατακτικά αποτελέσματα για το έτος 2009, κυρίως ε, για τον ερυθρό τόνο. Ε, το πρόγραμμα για το 2010 και 2011 τη νέα εντολή για την υπηρεσία μας βάσει του νέου κανονισμού ελέγχου που ανέκρινε πέρσι το Συμβούλιο και κάποιες καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Πρώτον, η αποστολή μας. Δύο είναι λέξεις κλειδιά. Ίση όρια ανταγωνισμού, level playing field και δεύτερον ε, η συμμόρφωση. Όσοι ασχολούνται εδώ και καιρό με το θέμα της αλληλείας θα γνωρίζουν ότι είναι εκ των όνου κάνευ ίση όρια ανταγωνισμού, ούτως ώστε οι αλληλείς να έχουν ίσες ευκαιρίες, να την χάνουν της ε, ισότιμης μεταχείρισης. Είναι απαραίτητο για τη σωστή εφαρμογή της ΚΑΠ να θεωρούν ότι δεν υφίστανται διακριτική μεταχείριση οι αλληλείς. Επίσης, εκ των είναι να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα συμμόρφωση προς τους κανόνες. Αυτό συμβάλλει στους, στους ίσους όρους ανταγωνισμού. Θέλουμε οι αλληλείς να αποκτήσουν αυτή την οτροπία συμμόρφωσης και σε συνδυασμό με τις εθνικές αρχές έχουμε υψηλά κοινά πρότυπα για την εφαρμογή της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας έχει εγκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική που διέπεται από αυτόν τον νέο κανονισμό ελέγχων και τον νέο κανονισμό για την ε, λαθρέα και άνερχη ε, αλία που, που θα εγκριθεί στη συνέχεια και θα ε, λάβουμε υπόψη στη συνέχεια την ε, μεταρρύθμιση της κοινής ελευτικής πολιτικής που έχει προβλεφθεί για το 2012. Ε, Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους ειδικούς, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες για τους ελέγχους και θέλουμε να αναβαθμίσουμε την εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής εγκρίνεται ένα ετήσιο ε, πρόγραμμα εργασίας ε, και ακολουθούμε δύο στρατηγικούς άξονες. Ε, επιχειρησιακός συντονισμός μέσω των κοινών προγραμμάτων ανάπτυξης και ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων. Το πολιετές πρόγραμμα για τις δραστηριότητες μας υπάρχει εδώ σε ένα πίνακα, είναι λίγο περίπλοκο. Θα σας μοιράσουμε την παρουσίαση. Στη συνέχεια, μην ανησυχείτε. Έχουμε συνεργασία και συντονισμό για να κάνουμε ε, κοινέ αναλύσεις κινδύνου από κοινού με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Και θα οργανώσουμε τα εθνικά προγράμματα επί τη βάση της κοινή ανάλυσης κινδύνου. Ετησίως θα εκτιμούμε δε την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων. Σας είπα ότι έχουμε και ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων. Δηλαδή τι κάνουμε, εκπαιδεύουμε τους εθνικούς επιθεωρητές, δημιουργούμε τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση των δεδομένων και για τον κανονισμό για την αναρχιαλία θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες. Και όλα αυτά θα συμβάλλουν στην ε, προώθηση ε, ε, της συμμόρφωσης ούτω ώστε με ομοιόμορφο τρόπο να εφαρμόζεται η κοινή αλλιευτική πολιτική. Of Τώρα, συντονισμός των κοινών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Θέλ, επιθυμούμε να επιτύχουμε επιχειρησιακό συντονισμό. Ποιο είναι ο στόχο αυτών των προγραμμάτων. Τα ε, κράτη-μέλη θα έχουν τα ε, σκάφη τους και τα αεροσκάφη που θα υπάγονται ε, σε αυτά τα προγράμματα και θα γίνει κοινή ανάλυση κινδύνου για να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτού του εθνικούς πόρους σε συνδυασμό πάντοτε με του εθνικού εμπειρογνώμονε. Θα χρησιμοποιήσουμε επιθεωρητές από διάφορα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των προγραμμάτων ελέγχων για να πατάξουμε τη μη συμμόρφωση. Προσπαθούμε να ενεργούμε με ομοιόμορφο τρόπο, ούτω ώστε όλε οι επιθεωρήσεις που γίνονται βάσει ενό κοινού προγράμματο να επιτελούνται ομοιόμορφα και αντικειμενικά. Αν υπάρξει ε, παραβίαση, γίνεται η καταγγελία, συλλέγονται τα δεδομένα, όλα αυτά με αντικειμενικό τρόπο. Η λειτουργία του προγράμματος βασίζεται ε, στο πρόγραμμα ελέγχου και επιθεωρήσεων που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εκεί υπάρχουν και ορόσημα και προτεραιότητες και κοινά κριτήρια μέσα από αυτό το πρόγραμμα υλοποιούμε το πρόγραμμα ελέγχων και επιθεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και προκατακτικά αποτελέσματα από τα προγράμματα για το 2009. Θα πλήξετε, θα σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία, αλλά τι να κάνουμε. Ε, στη Βαλτική, στη ΕΑΦ, στη ΝΑΦΚΟ έχουμε δραστηριοποιηθεί σε όλες αυτές τις περιοχές Έχουμε κάνει πολλές ημέρες επιθεωρήσεων. Ημέρες στη θάλασσα για την επιθεώρηση αλλά υπήρχαν και επιθεωρήσεις στους λιμένες Βλέπετε πόσα σκάφη περιπολίας είχαμε, τα αεροσκάφη, μικτές ομάδες επιθεωρητών, μικτές έτσι γιατί προέρχονται από διάφορα κράτη-μέλη, αριθμός ε, επιθεωρήσεων, ε, πολύ ε, υψηλό αριθμό στη Βαλτική, παραδείγματο χάρη. Στην Αύκο κυρίως στη θάλασσα γίνονται οι επιθεωρήσεις. Ε, λιγότερες επιθεωρήσεις γίνονται για τις εκφορτώσεις. Βλέπετε και τον αριθμό των παραβιάσεων ε, που ε, τεκμηριώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. Then we have Το θέμα του γαλαζόπτερου τόνου βλέπετε εδώ, αν τον βλέπετε βέβαια, τον αριθμό των περιπολούντων σκαφών. Υπάρχει και ο αριθμός των περιπολούντων αεροσκαφών στις περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά έχουν καθοριστεί μέσα στο κοινό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο έχει καθορίσει ο φορέας μας και φυσικά είναι πολλαπλές και πολυσχητήσεις δραστηριότητές μας για να εξασφαλίσουμε ότι ο γαλαζόπτερος αλλά ερυθρός τόνος ελέγχεται με τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την νομοθεσία μας. Οι κύριες δραστηριότητες έχουν λάβει χώρα στο κύριο μέρος της σεζόν, αλλά έχουμε καλύψει όλο το χρόνο, όλες επίσης τις περιοχές οι οποίες εμπλέκονται ιδίως στο φθινόπωρο στον Ανατολικό Ατλαντικό. Οι δραστηριότητες με το 2009 για τον γαλαζόπτερο τόνο είχαμε περίπου 74 παραβιάσεις όλες έτυχαν κοινοποίησης προς την ICAT και συζητήθηκαν εκεί στη συνάντηση της ICAT που έλαβε χώρα στο τέλος του 2009. Ενσωματώσαμε όλες τις πληροφορίες του φορέα μας σε μια έκθεση η οποία έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ICAT. Βλέπετε μια διαφάνεια για τις φαινομενικές παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τον γαλαζόπτερο ή ερθροτόνο <clears throat> και βλέπετε επίσης ότι χωρίζουμε αυτά τα πλοία τα οποία έκαναν τις παραβιάσεις ή παραβάσεις σε κοινοτικά πλοία και σε πλοία τρίτων χωρών. Σε ό,τι αφορά για τα προγράμματά μας μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα ότι βελτιώθηκε το 2009 σημαντικά η παρακολούθηση και η εποπτεία της αλίας του ερυθρού τόνου. Αυτό έχει επικυρωθεί από όλους και από την ΑΙΚΑΤ επίσης και ο συντονισμός από τον φορέα μας της ανάπτυξης μέσων εποπτείας και ελέγχου και ανταλλαγή επιθεωρητών μεταξύ 100 μελών ή το αξιοσημείωτος ή το πολύ αποτελεσματική και η ανάλυση κινδύνου περαιτέρω. Και οι περισσότερες παραβιάσεις είχαν να κάνουν με την ελλειπή τεκμηρίωση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις στατιστικές, ε, τα στατιστικά έγγραφα και τις δηλώσεις μεταφοράς. Αυτό ήταν ε, το συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε από μια εκστρατεία που ήταν μια κοινοτική εκστρατεία. Είχαμε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους. Πιστεύω λοιπόν κυρία Πρόεδρε και Αναφέρομαι στον κύριο Στίβενσον, ο οποίος ήταν επίσης παρόν εδώ το 2007, όταν έχουμε κάνει μια ακρόαση με τους αλείς ερυθρού τόνου. Το 2007 ήταν αρκετά χαοτικά τα πράγματα ακόμα, αλλά <clears throat> εμείς κάναμε τις προσπάθειες, θα επερχόμε τα επόμενα έτη για να ελέγξουμε και να εφαρμόσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την αλία του ερυθρού τόνου θέλω να αναφέρω λιγάκι και ορισμένα πράγματα για τον προπολογισμό του φορέα μας. Γιατί έχουμε προπολογισμό. Έχουμε. Είναι κυρίω διοικητικέ δαπάνε, δηλαδή κυρίως μισθοδοσία. Και υπάρχει και ένα τμήμα αυτού του προπολογισμού που αφορά τι λειτουργικέ δαπάνε. Είναι το γαλάζιο κομμάτι καμία σχέση με το χρώμα του φτερού του τόνου, περίπου 1,4 εκατομμύρια το 2010. Αυτά είναι τα ποσά που χρησιμοποιούμε για τις λειτουργίες μας δραστηριότητες. Για το <clears throat> πρόγραμμα εργασία μας, του 2010 και 2011, για τα δύο αυτά χρόνια θα βασιστούμε στα κεκτημένα των προηγουμένων ετών στα τρία πρώτα χρόνια της ε, λειτουργίας του φορέα μας. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες μας ξεκίνησαν το 2007. Έχουμε μια φιλοδοξία να ανταποκριθούμε στο νέο κανονισμό ελέγχου. Για να γίνει αυτό πρέπει ο φορέας μας να δουλέψει με πλήρη ικανότητα τα επόμενα χρόνια, με το, όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Η στρατηγική μα να υποστηρίξουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική και την μεσοπρόθεσμη στρατηγική που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Αλίας. Πρέπει επίση να ορθολογικοποιήσουμε ω το βαθμό του δυνατού τις ενέργειέ μα για να εκμεταλλευτούμε στα, στο έπακρο του περιορισμένου χρηματοοικονομικούς πόρου μα και γι' αυτό το λόγο έχουμε υιοθετήσει μια σειρά από προτεραιότητε για τον ρόλο του φορέα μα το 2010 και το 2011. Οι προτεραιότητε λοιπόν για το 2010 και το 2011 είναι κυρίω η νέα προτεραιότητα, είναι η άναρχη και ελαφραία αλία. Έχουμε στο φορέα μας μια σειρά από καθήκοντα στα πλαίσια του κανονισμού IUU, δηλαδή ανέρχης και λαθρέας Αλίες. κυρίως τα προγράμματα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των αλλιευμάτων βάσει των προγραμμάτων ειδικού ελέγχου και παρακολούθησης. Θα προσπαθήσουμε να μην είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί και θα αναπτύξουμε και την δημιουργία ικανότητας, δηλαδή κατάρτιση για τους εθνικούς επιθεωρητής αλίες συμβάλλουν έτσι στο να υπάρξει καλύτερη ε, συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών. Όπως ξέρετε, η ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε το 2007, περιείχε πολλές επικρίσεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο είχαμε αντιμετωπίσει τη συλλογή πληροφοριών βάσει της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ιδίως τις πληροφορίες ελεκτικού χαρακτήρα ο λειτουργικός συντονισμός. Έχουμε ένα προϋπολογισμό για το 2010 συνολικά 846.000 ευρώ. Θα έχουμε τέσσερα κοινά σχέδια ανάπτυξης και θα εργαστούμε και για τη λαθρέα και άναρχη αλληλεία. Θα διευρύνουμε το, την εμβέλεια των προσπαθειών μας, ιδίως για τον <clears throat> ερυθρό τόνο, τη λαθρέα και αναρχή αλληλεία. Θα εδραιώσουμε τα προγράμματα ανάπτυξής μας ιδίως για τον γάδο της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας και θα επεκτείνουμε και την ανάλυση κινδύνου σε ό,τι αφορά τα πολυετή προγράμματα αυτού του είδους και θα έχουμε μια κοινή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των τελευταίων προγραμμάτων. Το νέο κοινωτικό σύστημα για τον αγώνα κατά της IUU, της Λαθρέας και Αναρχισαλίας, αναφέρεται στην ε, ανακοίνωση της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη στους περιφερειακές, στους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης της ε, αλίας, άρνηση εκφόρτωσης ε, ή μεταφόρτωσης αλλιευμάτων, εφαρμογή της πιστοποίησης, πληροφορίες για την ε, πολιτική αυτή και ε, εκθέσεις ατενήσεως παρανομής αλίας. Έχουμε λοιπόν και ελέγχους σε τρίτες χώρες αιτήσει τη Κομισιόν και επίσης εκπαίδευση <clears throat> κοινοτικών επιθεωρητών και επιθεωρητών από τρίτε χώρες. Ό,τι αφορά τον ερυθρό τόνο για το 2010, τα κύρια στοιχεία είναι ότι θα έχουμε μια χάρτα Συγγνώμη, θα έχουμε ένα πλοίο το οποίο θα αναβλώσουμε, <clears throat> το οποίο είναι το ίδιο σκάφο το οποίο χρησιμοποιεί τώρα στην, στον, στην περιοχή Νάφο στον βορειοδυτικό Ατλαντικό, το πλοίο αυτό θα λειτουργεί με κοινοτική σημαία και στην Μεσόγειο ως ένα ουδέτερο σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα το χειρίζεται ο φορέας μας για ένα μήνα περίπου και θα χρησιμοποιήσουμε το σκάφος αυτό για να προσφέρουμε και συνεργασία σε τρίτες χώρες κράτη που δεν βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή της Μεσογείου και επίσης για την εκπαίδευση επιθεωρητών και για την εκτέλεση επιθεωρήσεων. Θα προσπαθήσουμε επίσης μαζί με την Κομισιόν να φέρουμε σε πέρας μια σειρά από ε, επιθεωρήσεις σε ξένα νερά, νερά άλλων κρατών μελών τη Μεσογείου. Θα υπάρξει και μια πλατφόρμα συντονισμού που θα αναπτυχθεί από τον φορέα μας στο Βίγο με συμμετοχή των κρατών μελών με έδρα στο Βίγο <clears throat> και θα συντονίσουμε αυτή την συνολική δραστηριότητα με πλοία αεροπλάνα. Θα υπάρξει ο συντονισμό από το Βίγο και σε καθημερινή βάση θα έχουμε πληροφορίες από τις ομάδες επιθεώρησης. Αναλύουν εμείς όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες θα βασίζονται σε πρώτερο κίνδυνο, μάλλον ανάλυση, πρώτερη ανάλυση κινδύνου και θα εστιάσουμε τις δραστηριότητές μας στην ε, ανείχνευση πρακτικών οι οποίες δεν είναι σύμμορφες με τους κανονισμούς για την αλία του ερυθρού τόνου. Και πάλι θέλουμε να εκπαιδεύσουμε και να καταρτήσουμε επιθεωρητές από όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό το κάναμε και το 2008 και θέλουμε να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της κατάθεσης, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που μπορεί να προκύψει στο έργο αυτών των επιθεωρητών. Για την κατάρτιση έχουμε ένα προϋπολογισμό 564.000 ευρώ. Θα υποστηρίξουμε την υποδομή ελέγχου και παρακολούθησης, την παρακολούθηση των δεδομένων, τις κοινέ ικανότητες και μια πλατφόρμα συντονισμού για αυτές τις ενέργειες και επίσης θα αναπτύξουμε το ανθρώπινο δυναμικό με συντονισμό της εκπαίδευσης επιθεωρητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. το ταχύτερο δυνατό. Θα πάρουμε τη νέα αυτή, θα εγκρίνουμε αυτή τη νέα οδηγία για τον φορέα μας βάσει του κανονισμού ελέγχου. Υπάρχουν κάποια σημαντικά, σημαντικά θέματα. Το προσωπικό μας θα έχει το χαρακτήρα των επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή νερά. Έχουμε τις εξουσίες για να κάνουμε επιθεωρήσεις σε διεθνή ε, ύδατα με το συντονισμό του φορέα μας και έχουμε επίσης τη δυνατότητα να έχουμε και τα δικά μας μέσα για τις επιθεωρήσεις. Και αυτό υπάρχει και στη σχετική διάταξη στο νέο κανονισμό ελέγχου. Τα τελευταία χρόνια ε, ναυλώναμε σκάφη της ΝΑΦΟ και ναυλώσαμε και ένα σκάφος το οποίο χρησιμοποίησαμε φέτος το καλοκαίρι για τον ερυθρό τόνο και αυτό το χρηματοδότησαν τα κράτη-μέλη. Ο νέος ελεγκτικός κανονισμός μας επιτρέπει να χρωματοδοτούμε αυτά τα μέσα επί τη βάση του κοινοτικού προπολογισμού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα στις ε, δημοσιονομικές ε, πολιτικές προοπτικές ε, πρόβλεψη για χρηματοδότηση στα σκάφη αυτά και θα κάνουμε το ίδιο που κάναμε και το 2010, χρηματοδότηση δηλαδή από τα κράτη-μέλη για το 2011. Από εκεί και πέρα λογικά θα πρέπει να έχουμε χρηματοδότηση από τον κοινοτικό ε, προϋπολογισμό και ε, θα πρέπει να γίνει χρηματοδότηση για να γίνουν αυτά και το 2011. Η νέα δυνατότητα που έχουμε στο νέο ελεγκτικό κανονισμό είναι να υπάρχει και μία ομάδα εκτάκτου ανάγκης. Έχουμε προβλέψει λοιπόν να υπάρχει μια μονάδα, ένα τμήμα εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που χρειάζεται άμεση επέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο και ε, η υπηρεσία θα είναι σε θέση να κάνει αυτή τη δουλειά, να συντονίσει τις δραστηριότητες ε, μέσω αυτής της μονάδας εκτάκτου ανάγκης. Κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ε, ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας το 2007 και επομένως έχουμε ελάχιστο προσωπικό. Έχουμε 8 επίσημους επιθεωρητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ξεκινήσαμε τις επιχειρήσεις μας το 2007. Φέτος θα είμαστε περίπου 60 άτομα στην υπηρεσία και ε, ανυπομονούμε ιδιαίτερα να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξε μεγαλύτερη συνεργασία στα κράτη-μέλη από ό,τι στο παρελθόν, κυρίως ε, σε θέματα στα οποία διαδραστηριοποιείται ο οργανισμός μας. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη στις διευθυντικές ομάδες και γίνεται ένας συντονισμός στις λεγόμενες κοινέ τεχνικές ομάδες ε, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτές οι επιχειρήσεις γίνονται ε, στα πλαίσια κοινοτικών προγραμμάτων. Ε, στα πλαίσια της συνεργασίας μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η συνεργασία ήταν περισσότερη από ό,τι ποτέ άλλοτε την τελευταία τριετία χάρη στη δημιουργία του οργανισμού μας. Επίσης, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων βελτιώθηκε. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και να πούμε ότι στα πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της, του οργανισμού θα γίνει μία αναθεώρηση ε, και θα πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση για να εξαγάγουμε συμπεράσματα για την προστιθέμενη αξία της υπηρεσίας. Νομίζω ότι ήδη από σήμερα όμως μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ε, είχαμε τα θέματα του ερυθρού τόνου, το γάδο στη Βαλτική θάλασσα και όλα αυτά βελτιώθηκαν χάρη στην ενισχυμένη συνεργασία των εθνικών αρχών των ε, κρατών μελών η οποία συντονίστηκε από την υπηρεσία. Θεωρούμε ότι ε, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά έχει γίνει μια πρώτη συνεισφορά ε, ώστε να είναι ισότιμο το πεδίο για όλους τους αλλιείς, για όλη την αλλιευτική ε, δραστηριότητα και όλο τον κλάδο και πήραμε και πολλές θετικές απαντήσεις από τους αλλιες καποια Κάποια κράτη-μέλη ε, επιθεωρήθηκαν και από επιθεωρητές από τη χώρα τους και χάρηκαν που υπήρχε μια ίση μεταχείριση σε αυτή την περίπτωση και γνώριζαν ότι οι αλληλεί ε, τη χάνουν τη ίδια μεταχείρισης όταν αλλιεύουν το ίδιο είδο όταν έχουμε αυτό το κοινό σχέδιο ε, Είμαστε στη διάθεσή σας ε, για την ε, Επιτροπή ε, Αλληλείας. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να βελτιωθεί η κοινή αλληλευτική πολιτική και όσον αφορά στη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι μία από τις αδυναμίες της κοινής αλληλευτικής πολιτικής ήταν το θέμα της εφαρμογής της. Σε κοινωτικό επίπεδο λοιπόν θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική αυτή εφαρμόζεται καταλήλως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστερ. Θα δώσω το λόγο στους βουλευτές οι οποίοι ζήτησαν το λόγο. Κύριος Εστίδων, στον πρώτο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κώστερ. Είναι πολύ θετική η έκθεση που μας παρουσιάσατε και προσβλέπω στο να έλθω μία μέρα στο όμορφο Βίγο να παρουσιάσω να, να δω το κέντρο που μας παρουσιάσατε και προτού δημιουργηθεί αυτό το κέντρο τα πράγματα ήταν αρκετά χαοτικά και εμείς ακούγαμε πάντα από τους ψαράδες μας, τα δικά μας κάτι μέλη ότι <clears throat> τα δικά μας κράτη-μέλη είχαν 10 φορές περισσότερους επιθεωρητές από ό,τι τα άλλα κράτη-μέλη. Φυσικά επιλύθηκε αυτό το πρόβλημα με το φορέα του Βίγο. Υπάρχει ακόμα ένα εκκρεμές πρόβλημα το οποίο οδηγεί σε έλλειψη ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των αλλιέων και ίσως θα μπορούσατε να θίξετε και αυτό το θέμα ενώπιον των κρατών μελών και εσείς έχετε το έργο του ελέγχου και της επιθεώρησης. Εγώ αναφέρομαι όμως εδώ στο δικαστικό σύστημα των κρατών μελών και τις κυρώσεις που επιβάλλονται γιατί για παρά, παρόμοια αδικήματα σε διαφορετικά κράτη-μέλη υπάρχουν τελείως διαφορετικές ποινές που επιβάλλονται. Και πέρσι είχαμε μια υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου μια ομάδα που ήταν πατέρας και γιος αλής στη Σκοτία κατηγορήθηκαν ότι εκφόρτωσαν παράνομα γάδο. Τους καταδικάσανε να πληρώσουν χίλιες λίρες, μόνο 700 καταφέρανε να βρουν με, θέτοντας τα σπίτια τους σε υποθήκες και μπήκαν και δύο φυλακοί λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση. Εγώ δεν θέλω να συγχωρήσω την παράνομη αλία για, ένα παρόνυμο, παρά, την παράνομη ε, εκφόρτωση σε ένα κράτος μέλος δεν θα είχαν να πληρώσουν τέτοιο πρόστιμο. Αν δεν μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε αυτό το επίπεδο ισότιμου ανταγωνισμού και στις ποινές, αν, έχουμε τις ίδιες, αν δεν έχουμε τις ίδιες ποινές, θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τους αλληλείς ότι υπάρχει πραγματικά ίση μεταχείριση για όλους τους αλληλείς. Μακρά εμού ως Βρετανού συντηρητικού να ζητήσω να υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση σε ό,τι αφορά τις δικαστικές ποινές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα με διώχνανε από το κόμμα μου αύριο. Αλλά τουλάχιστον θα μπορούσατε να κάνετε προτάσεις προς τα κάτι μέλη <clears throat> ότι εφόσον έχετε επιτύχει αυτό το οποίο σίγουρα φαίνεται να έχετε επιτύχει στο καθεστώς της εποπτείας και επιθεώρησης, τα κάτι μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να συντονίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την επιβολή ποινών. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο, στους βουλευτές πάλι. Ο κύριος Ρωμέβα, ευχαριστώ πάρα πολύ Χαίρομαι που βελτιώνεται η κατάσταση τόσο σε ό,τι αφορά την επιμελητία και στην αντιμετώπιση αυτών των δραστηριοτήτων. Δύο ερωτήματα. Ένα είναι πολύ πρακτικό. Κατά την άποψή σα, ποια είναι η καλύτερη στιγμή να έρθουμε στο Βίγο σε ό,τι αφορά τα δραστηριότητά σα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε στιγμέ που έχετε ειδικά καθήκοντα τα οποία είναι ενδιαφέρον να τα δούμε και σε άλλε εποχέ είναι πιο νεκρή περίοδος. Ποια είναι η καλύτερη εποχή κατά την άποψή σας να έρθουμε να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις στο Δίκτυο. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το ουσιαστικότερο ερώτημα για τον ερυθρό τόνο. Οι παρατηρήσεις μου καταρχήν αναφέρονται στα στοιχεία τα οποία μας δώσετε. Αναφερθήκατε στις, στις φαινομενικές παραβάσεις. Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ αυτών των φαινομενικών παραβάσεων και των παραβάσεων που έχουν πράγματι διαπιστωθεί και έχουν τύχει συνέχειες. Και δεύτερον, πώς θα διευρύνετε την εμβέλεια των ενεργειών σας για τον ε, ερυθρό τόνο, όπως είπατε, και το νέο κείμενο το οποίο έχει εγκριθεί παρέχει κάποιες ευκαιρίες να λύσουμε τα προβλήματα δεδομένων. Ποια είναι η σύστασή σας στο θέμα αυτό. Και τέλος έχω μια πολιτικού χαρακτήρα ερώτηση. Υπάρχει πια ένας κίνδυνος, κάτι το οποίο μας έχουν πει πολλές φορές, ότι λόγω της μείωσης των ποσοστώσεων για τον ερυθρό τόνο θα αυξηθούν οι παραβιάσεις, οι παραβάσεις και οι παράνομοι αλίευ. Αυτό έχει αναφερθεί ότι θα γίνει στην Ιταλία και σε άλλα μέρη. Επίσης, μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένο, αν εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο κίνδυνος και δεύτερον, αν αυτό είναι κάτι που θεωρείτε ότι είναι πιθανό να συμβεί, ποια θα είναι η απάντηση που μπορεί ο φορέας του Βίγο να αναλάβει για να υπάρξει έλεγχος. Η κυρία Λεβίν τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ για την παρακολούθηση των αλλιευμάτων ερυθρού τόνου. 1,4 εκατομμύρια ευρώ νομίζω είναι το κονδύλι που αναφέρατε για την παρακολούθηση. Αυτό αντιστοιχεί στο προπολογισμό της υπηρεσίας αποκλειστικά ή και των κρατών μελών. Α, δικό σας προϋπολογισμός. Μάλιστα. Γιατί δεν φαίνεται και τόσο μεγάλο το ποστό. Είναι ευρεία εμβέλεια σε δραστηριότητα παρακολούθησης. Δεύτερη ερώτηση λοιπόν. Πόσο τι, ποιο ποσό θα χρειαζόταν για να έχουμε μια καλή παρακολούθηση για τον ερυθρό τόνο στο σύνολο της Μεσογείου. Ε, μια εκτίμηση μπορείτε να κάνετε σε ευρώ. Πόσο θα κόστιζε. Και για μία από τις διαφάνειες για τη Βαλτική θάλασσα που μας δείξατε φαίνεται να έγιναν πάρα πολλές ε, επιθεωρήσεις αλλά όχι και τόσες πολλές παραβάσεις. Ε, γιατί? οι αλληλείς της Βαλτικής ε, ε, είναι πιο νομοταγείς ή μήπως ε, δεν είναι ικανοποιητικές οι επιθεωρήσεις. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που είχα να σας θέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων για τη Βαλτική θάλασσα και τα αποθέματα του γάδου κρίνεται ότι θα ε, είναι σε καλή κατάσταση βάσει των αποτελεσμάτων άρχισαν να εφαρμόζονται διάφοροι κανονισμοί και ίσως αυτός είναι ο λόγος. Παραδείγματο χάρη από 110 στα 120 mm περάσαμε για το μέγεθος των ματιών, των δικτυών ή παραδείγματο χάρη αυξήσαμε το μέγεθος των ματιών σε άλλα ε, είδη δικτυών από 90 που ήταν και έτσι έχουμε λιγότερες απορρίψεις. Στη Δυτική Βαλτική έχουμε πρόβλημα με τη Ρέγκα. Ε, σημειώθηκε εκεί δραματική μείωση του αποθέματος. Το δίχτυ για την αλία της Ρέγκας έχει μέγεθος ματιού 32 mm και είναι δανέζικη γρήπη, ε, διατλαντική τεράστια τεράστια σκάφη ενώ το βάθος είναι μόνο 55 μέτρα στη Βαλτική και ψαρεύουν τα πάντα, τα σαρώνουν όλα αυτά τα τεράστια σκάφη και κανείς δεν λέει τίποτα, δεν ελέγχει κανείς ε, τα ε, αλλιεύματα στη Βαλτική και χρησιμοποιούνται για παραγωγή χθιαλεύρων ε, στη συνέχεια. Πώς ακριβώς ελέγχετε εσείς αυτήν την αλία, πώς ακριβώς ενεργεί η υπηρεσία σας για να καταπολεμήσει την αλία αυτών των σκαφών κατόπιν για τις ιστοσελίδες της υπηρεσία σας. Εξαφνικά εξαφανίστηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Για ποιο λόγο παρακαλούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω τον κύριο Κόσνερ και να σας ε, πω ότι εγώ ε, έτυχα εξαιρετικής υπεδοχής ε, στη Γαλλικία. Ο ρόλος της υπηρεσίας εκτιμάται όλο και περισσότερο και αξιολογείται πάντα καλύτερα. Η ερώτησή μου είναι το εξής, η εξής. Εάν ε, οι έλεγχοι φτάσουν στο 100% θα πρέπει να βρούμε, να κάνουμε μια διάγνωση ως προς τα ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Εσείς πού θα θέτατε έμφαση, ε, τι θα πρέπει να κάνουμε για να τα επιλύσουμε και το θέμα του τι γίνεται με την ε, καλλιέργεια και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λέτε ότι έχουμε περισσότερη συνεργασία στα κράτη-μέλη. Πώς θεωρείτε ότι εκλαμβάνεται ο ρόλο της υπηρεσίας. Θα ήθελα και εγώ να σας κάνω μια ερώτηση, λέει η Πρόεδρος. Καταρχάς, να πω ότι επειδή του χρόνου θα ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο να αρκεί ή όχι ο προπολογισμό της υπηρεσίας και αν θεωρείτε ότι πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό της. Δεύτερον, για το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Στο θέμα του ερυθρού τόνου, επί παραδείγματι, ε, αυτό που έχετε εσείς είναι μικρότερο από τη ΣΝΑΦΟ. Τι θέλω να πω, ότι όταν τα κονδύλια είναι λίγα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες και δεδομένα των προβλημάτων που έχουμε με τον ερυθρό τόνο και με τα όσα θα μπορούσαμε να έχουμε στο μέλλον με όλες αυτές τις συζητήσεις που είναι εξελίξεις, το πράγμα θα μπορούσε να φτάσει ε, στα χειρότερα. Επομένως, θα πρέπει ε, να δούμε κατά πόσο θα πρέπει εμείς να εστιάσουμε στον ερθρό τόνο περισσότερο από την άφο. Είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται ε, τόσο πολύ. Ε, υπάρχουν άλλα είδη που δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και ίσως θα έπρεπε να εστιάσουμε εκεί. Γιατί εσείς λοιπόν με τον, στον προϋπολογισμό σας δεν δίνετε ακόμα περισσότερη προτεραιότητα στον ερθρό τόνο που ξέρουμε ότι Εάν μπει στο παράρτημα ένα του site που είναι αυτό που εγώ θα επιθυμούσα, καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστούμε και περισσότερους ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον ε, το θέμα θα ελέγχεται και θα τηρούνται οι υποχρεώσεις και δεν θα εξαντληθεί το απόθεμα όπως ε, πιστεύουν κάποιοι. Τέλος, ε, να σας δώσω το λόγο, πάρτε όσο χρόνο θέλετε και απαντήστε σε όλα όσα σας ρώτησαν οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, Λεωπρό. Ο κύριος Κώσε. Το ερώτημα του κύριου Στίβενσον. Τι μπορούμε να κάνουμε και ποια είναι και η εντολή μας. Η εντολή μας φτάνει μονάχα μέχρι τις επιθεωρήσεις και τη